έργο και αυτό πρόκειται να βοηθήσει την ε, Ευρώπη και την κληρονομιά τη, διότι ε, ε, τώρα αποδείχθηκε ότι χωρί κανεί να δαπανίσει πολλά χρήματα μπορεί κανεί να έχει αυτή την προσθεθεμένη ευρωπαϊκή αξία. Και επίση πιστεύω ότι όπου αυτό το σήμα απονέμεται θα έχουμε μεγάλο κέρδος. Θα έχουμε πολύ περισσότερες ε, επισκέψεις, τουρισμό, κυκλοφορία και όλο αυτό είναι υπέρ της ευρωπαϊκής οικονομίας. Άρα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η πολιτιστική ταυτότητα της Ευρώπης θα αναδειχθεί και όλοι σε όλο τον κόσμο θα, ε, θα, θα, θα, λάβουν γνώση αυτού του γεγονότος αλλά είναι πάρα πολύ φασαρία και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Ευχαριστώ πολύ, Αντινόρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το σήμα Ευρωπαϊκής ε, Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι ουσιώδους ε, σημασίας για μία ήπειρο στην οποία βρίσκονται οι περισσότερες τοποθεσίες ε, με το σήμα της UNESCO. Αρχαιολογικοί χώροι, αστικοί χώροι που έχουν παίξει σημαντικότατο ρόλο στην, στον πολιτισμό της Ευρώπης. Το σήμα λοιπόν Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι σημαντικό για την Ευρώπη και είναι και επικοδομητικό για τον πολιτιστικό διάλογο Ελπίζομαι ότι αυτή η επιλογή θα κάνει καλό και στις επόμενες γενιές έτσι ώστε να ενωθούν οι επόμενες γενιές από άποψη πολιτιστική. Συγχαίροντας ε, την ε, ε, εισηγήτρια θα ήθελα να την συγχαρώ κιόλας για τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο διεύθυνε τις διαδικασίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε τώρα στην σύσταση της κυρίας Πακ για τη συμμετοχή Ελβετικής Ομοσπονδίας στο πρόγραμμα Νεολαία σε δράση και στο πρόγραμμα Δράση στον τομέα της μάθησης διαβίου. Ο κύριος Πάκουλα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω ότι η διαβίου ε, μάθηση γυράσκωνα ή διδασκόμενο είναι μια μεγάλη ευτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια ευκαιρία να ευχαριστήσω την Δόρη Σπάχ για τη θαυμάσια εργασία τη. Εγώ προφανώ υπερψήφιζα. Και πάνω απ' όλα δείχνει ότι οι ευρωσκεπτικιστές δεν έχουν δίκιο. Θέματα όπως η διαβίου μάθηση δεν είναι μονάχα μια μεγάλη επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά γνωρίζουμε ότι και χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η ακριτική Ελβετία ενδιαφέρονται και θέλουν να καταβάλουν χρήματα για να έχουν και αυτέ συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα. Με τέτοιο τρόπο μπορούμε να έχουμε ανταλλαγή βελτίστων πρακτικό και να κάνουμε τα προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ευρύτερα διαθέσιμα. Προγράμματα για τη νεότητα, προγράμματα για την ενεργό γύρανση. αυτά είναι προγράμματα πολύ θετικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να χαιρετήσω την είσοδο τη Ελβετία σε αυτά τα προγράμματα. Ευχαριστούμε πολύ. Χάναν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα <clears throat> στην Ολομέλεια. Γιατί η Ελβετία τα καταφέρνει τόσο καλά. Θα φανταζόσασταν ότι μια χώρα η οποία είναι ιδιαίτερα ε, τρωτή στην χρηματοοικονομική κρίση θα είχε θυγεί πάρα πολύ. Αλλά 214% ήταν το ΑΕΠ κατά κεφαλήν της Ελβετίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο φορές πιο πλούσιοι από τις πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά μέσο όρο. Αυτό δείχνει πόσο καλά έχουν συμφωνήσει οι Ελβετοί για, με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύπτονται από την ενιαία αγορά, αλλά είναι έξω από την πολιτική γεωργικών θεμάτων, από την αλληλεία, δεν πληρώνουν στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ρυθμίζουν μόνοι του τα θέματα ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουν την ευκαιρία να έχουν ελεύθερε συμφωνίε με όλε τι τρίτε χώρε. Αν μπορούν λοιπόν με τι διμερεί συμφωνίε οι Ελβετοί να έχουν το καλύτερο βιωτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο περισσότερο ένα ε, εμπορικό έθνο και θαλάσσιο έθνο όπω είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να πάρουμε πίσω την εξουσία μας, να έχουμε την τοπική δημοκρατία όπως και η Ελβετία και να μπορέσουμε να μειώσουμε την επαφή μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ελάχιστο. Ευχαριστώ. Eh, Περνάμε τώρα σε, στην έκθεση Σάγερ, έλεγχος από τα κράτη-μέλη της άρχης των εκτελεστικών αμοιωτήτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Μουσκαρντίνη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ απέσχον στη σημερινή ψηφοφορία, σε αυτή την έκθεση επιτροπολογίας, γιατί για μία ακόμα φορά γίνεται προσπάθεια να γίνει μη εφαρμοστέα ή να αφαιθεί ε, στην ε, ευχέρεια, στη διακριτική ευχέρεια των κρατών η εφαρμογή της ε, απαγόρευσης τρέβλωσης του ανταγωνισμού. Παρότι φτάσαμε σε μια συμβαστική λύση με το Συμβούλιο, Παρόλα αυτά λέγω δεν καταφέραμε να ευθυγραμμίσουμε τις εμπορικές πολιτικές με την επιτροπολογία κυρίως στο σκέλος των εμπορικών συναλλαγών που ιδιαιτέρως πλήττει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης όπου ε, κανόνας έχουν γίνει πλέον οι μετατοπίσεις ε, επιχειρήσεων και πλήττοντας έτσι σφοδρότατα την ευρωπαϊκή οικονομία. Ο κύριος Χανάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα σας το πω όσο πιο απλά μπορώ. Ε, στην ουσία έχουν επιβληθεί, έχει επιβληθεί ζυγός ε, στους ληστεύονται ε, οι ε, πολίτες και της Ευρώπης και της Ιρλανδίας έτσι ώστε να ξεπεραστεί η κρίση στο τραπεζικό σύστημα και Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δυνατόν να πεις ότι βοηθάς ένα χρεωμένο φίλο με το να του βάλεις το πιστόλι στον κρόταφο. Από το 1998 μέχρι το 2007 ε, τα επιτόκια ήταν μείον 1% στην ε, Ιρλανδία ε, και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γιατί δεν μπορούν να αυξήσουν τα επιτόκια και τώρα με την κρίση ακόμα λιγότερη περιθώριο κίνησης έχουν και επομένως ποια λύση έχουν να φύγουν από τις χώρες τους. Στην ουσία θα έπρεπε να βοηθήσουμε την Ιρλανδία έτσι ώστε να διασωθεί το ευρώ, να διασωθεί η, ε, η, κατάσταση στην ουσία και να, να βοηθηθεί η χώρα έτσι ώστε να ξεπληρώσει τα δάνειά της και όχι να της δώσουν μία να πάει ακόμα πιο βαθιά. Ευχαριστώ πολύ επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση Αντρίκεν για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και το 2009 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Πρέντα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πρώτα πρώτα να συγχαρώ την κυρία Αντρικένε διότι κατέβαλε προσπάθεια για αυτή την έκθεση. Εγώ ψήφισα για την τροπολογία 25 θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνος από το κλίμα στην Ρωσία. Θα πρέπει κράτος δικαίου, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα να τα υπερασπιζόμεθα. Όμως πάρα πολλοί ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα είχαν δράσει στη Ρωσία για το οποίο σημαίνει ότι όπως λέει η τροπολογία χρειάζεται να διερευνηθούν τα εγκλήματα βάρος των ακτιβιστών. Η πρωτοβουλία μας δείχνει ότι η Ρωσία παρακολουθεί το τι σχολιάζουμε εμείς για την κατάσταση εκεί και όμως θα πρέπει να συνεχιστεί ε, η παρακολούθηση των εξελίξεων εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Καλινόφσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πάντα τους ασθενέστερους αυτούς οι οποίοι αντιμετωπίσουν διακρίσεις, τους φτωχούς και αυτούς που έχουν ανάγκη βοήθεια σε όλο τον κόσμο. Εμείς δίνουμε το βραβείο Σαχάροφ, το απονέμουμε <clears throat> κάθε χρόνο. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλάκις δεν εφαρμόζει στο έδαφος της το σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα να καταδείξω ποια είναι η διάκριση που υπάρχει εναντίον μειονοτήτων παραδείγματο χάρη τη πολωνική μειονότητα στη Λιθουανία, παρά τι διεθνεί συμβάσει για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι χάνουν ακόμα διακρίσεων. Η Λιθουανία αυτή τη στιγμή περιορίζει την ε, εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα για τις μειονότητες στην Λιθουανία. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τα ανθρώπινα δικαιώματα την χάνουν σεβασμού στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκής η μείωση της εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα, το κλείσιμο των πολωνικών σχολείων είναι σαφώς μια διακριτική μεταχείριση αυτής της μειονότητας. Grazie, la parola all'onorevole Kelam. Kelam. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ υποστήριξα την τροπολογία υπαριθμών 25, ιδιαίτερα το δεύτερο τμήμα της, διότι θεωρώ ότι είναι ζωτικού χαρακτήρα. Λέει το τμήμα αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να σκεφτεί να απαγορεύσει την είσοδο Ρώσων αξιωματούχων που έχουν να κάνουν με περιπτώσεις ε, δίωξης και δολοφονίας ε, αντιφρονούντων και επίσης να εξασφαλίσει το πάγωμα των στοιχείων ενεργητικού αυτών των ατόμων σε όλα τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και για τη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω να ενθαρρύνω ιδιαίτερα και να παρατρύνω την Κομισιόν και το Συμβούλιο να ακολουθήσουν αυτή την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουν αυξηθεί οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρόσφατα. Τώρα θα πρέπει να σταματήσουμε απλώς να διαμαρτυρόμαστε και θα πρέπει να δράσουμε, να δημιουργήσουμε πραγματικά προβλήματα σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η συνεργασία της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει πραγματική προοπτική αν ο Μαγρέτσκι, οι, οι περιπτώση Μαγρέτσκι και Χοδωρόφσκι αντιμετωπιστούν σωστά από τα δικαστήρια και οι υπεύθυνοι για όλα αυτά τα κακά να τιμωρηθούν. Κυρία Πρόεδρε, εγώ ψήφισα υπέρ της έκθεσης Αντρική Ένα. Είναι σημαντικό το να τίθενται τέτοια θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως πάντα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και στην πράξη ενεργούμε σύμφωνα με όσα διακηρύσουμε. Δεν είναι πάντα εύκολο αυτό βέβαια. Πώ θα το κάνουμε όμω. Ίσως θα έπρεπε να έχω υποβάλει ένα διαδικαστικό. Όταν συζητήθηκε η έκθεση Ελάκη. 50 ήταν εκείνοι που σηκώθηκαν. 50 μας είπαν ότι είναι 40 μετά. και νομίζω θα πρέπει να τηρούμε του κανονισμού γιατί δεν είναι εδώ. Όταν δεν μπορούμε να τηρήσουμε τα όσα προβλέπονται εδώ, δεν μπορούμε να λέμε στου άλλου τι να κάνουμε. Θα πρέπει επομένω να ενεργούμε σύμφωνα με νόμου και κανόνε και να σεβόμαστε και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν νομίζω επομένω ότι μπορούμε ακόμα να καταβάλουμε προσπάθεια για να αποκτήσουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία και μετά να καθόμαστε και να α, προτείνουμε στο τι θα κάνει και η Ρωσία και οι άλλοι. Βεβαίως και θα πρέπει να καταπιέζονται οι μειονότητες, όλοι θα πρέπει να απολάβουν αυτών των δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση Αρλάκη. Νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν. Και θα δώσω τον λόγο στον κύριο Βαν Τάλεν. Eh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δείξει και πάλι σε ποια, ποια πλευρά υποστηρίζει η Αμερική έχει αποτύχει στο Αφγανιστάν και το η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιδράσει και να ξεκινήσει κάποιες πρωτοβουλίες. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι αν την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα πάνε καλά. Αν διαβάσει κανείς την συμφωνία ζητούμε <clears throat> την, ε, το ψήφισμα, ζητούμε από το Ιράν να συμμετάσχει στην ε, επίλυση των προβλημάτων στο Αφγανιστάν. <clears throat> Αλλά εγώ δεν μπορώ να δεχτώ κάτι τέτοιο, ότι ζητούμε από το Ιράν βοήθεια στα θέματα αυτά. Κάνουμε μια συμφωνία με το διάβολο. Εγώ είμαι 100% εναντίον μιας τέτοιας άποψης και αυτό καταψήφισα και την έκθεση. Κύριο Χάναν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είχα την τιμή να είμαι στο Αφγανιστάν με τις Βρετανικές δυνάμεις πρόσφατα στην αρχή του χρόνου. Όχι μονάχα συνάντησα οι Βρετανούς στρατιώτες, αλλά, και Δανούς και Εστονούς στρατιώτες. Πρέπει να πω ότι δεν μπορώ να εκφράσω αρκετά την ευγνωμοσύνη μου σε όλους αυτούς τους συμμάχους μας που έχουν κάνει προσπάθειες και τους υπερπόντιους συμμάχους μας φυσικά για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτής της δυστυχισμένης αλλά τόσο έμορφης χώρας. Θέλω να τονίσω ότι φαίνεται ότι κάνουμε ένα σφάλμα ως Δυτική Συμμαχία που έχει να κάνει με την πολιτική μας σε σχέση με την ε, εκρίζωση του, της καλλιεργίας του οποίου. Όλοι αυτοί οι οποίοι ξέρουν ε, για γεωργία ξέρουν ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο συντηρητικό από ένα μικρό γεωργό. Αλλά με την ε, άποψη αυτή ότι πρέπει να εκκριζώσουμε τις καλλιέργειες του οποίου έχουμε κάνει όλους αυτούς τους καλλιεργητές να είναι αντίπαλοι μας λόγω της ε, ε, πολιτικής μας να καταστρέψουμε μια παραγωγή η οποία έχει παγκόσμια ε, ζήτηση. Υπάρχει ζήτηση οποίου για μορφήνη σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν επαναφέρουμε αυτή την καλλιέργεια θα δημιουργήσουμε τις βάσεις για μια ανθούσα με παπαρούνια άνθη κοινωνίας και οικονομίας στο Αφγανιστάν. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων για να διασφαλίζεται η χρηματοοικονομική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ ψήφου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα το σχετικό ψήφισμα όσον αφορά το μηχανισμό αντιμετώπιση των κρίσεων. Γιατί σε Ελλανδία και σε Ελλάδα βλέπουμε τι γίνεται στην πραγματικότητα, τι γίνεται με αυτούς τους μηχανισμούς που θέλουν να σώσουν δίθεν σύστημα. Ενώ οι κερδοσκόποι ε, το, μόνο το οποίο κάνουν είναι να προσπαθούν να, βγάλουν λεφτά εις βάρος των πιο φτωχών. Σήμερα, μάλλον θα αποφασίσει το Συμβούλιο να τροποποιήσει τη της Λισαβόνας και να έχει περισσότερες εξουσίες τόσο ώστε να επιβάλλει τους ε, όρους υπό τους οποίους θα δίνεται αυτή η, η αρρωγή σε, σε, σε κράτη-μέλη. Η Ιρλανδική κυβέρνηση δεν θα πρέπει να δεχθεί χωρίς δημοψήφισμα να εφαρμόσει τη νέα συνθήκη. Ε, προτεκτοράτο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου καταντήσαμε. Επομένω, απαιτούμε δημοψήφισμα για οποιαδήποτε αλλαγή τη συνθήκη τη Λισαβόνα. και έτσι ο λαός της Ιρλανδίας να έχει την ευκαιρία να πει το όχι όσον αφορά αυτή την κυριαρχία των αγορών. Ευχαριστώ πολύ. Ε, λύεται η συνεδρίαση μέχρι τις 15.00. Ε,